Και θα ήθελα να σας πω πως το σημείο 12 θα το δούμε αμέσως μετά το σημείο 10. Μετά. Περνάμε σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης. Ε, ανακοινώσεις του Προέδρου, αν δεν έχετε αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, ανακοινώσεις του Προέδρου. Να πω πως ε, είχαμε μια αλλαγή στον ε, κανονισμό. Και όταν υπάρχει μια προφορική τροπολογία, χρειάζεται τώρα πλέον το 5% των βουλευτών για να φέρουν αντίρρηση. Αυτή τη στιγμή επαρκεί ένας Τώρα το όριο είναι το 5% το οποίο στην Επιτροπή μας αντιστοιχεί σε δύο βουλευτές. Αν δεν φέρουν δύο βουλευτές αντίρρηση ε, μπορεί να προχωρήσει η προφορική τροπολογία. Σημείο 3. Τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων δεν είχαμε κάποια σχόλια, οπότε θεωρείται ότι εγκρίθηκαν. Το ίδιο και για το 4. Μετά έχουμε το σημείο 5, ψηφοφορία. Λοιπόν, σιγά σιγά θα κάνουμε την ψηφοφορία γιατί ξέρω πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πρέπει να μπορείτε να παρακολουθείτε. Ε, οπότε θα δώσω τον λόγο λοιπόν στην κυρία Παπαδοπούλου πρώτα απ' όλα. Thank you very much, ε, ε, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια έκθεση για τη φιλοκτονία αυτή εδώ. Η φιλοκτονία δεν έχει κάποιον ε, τυποποιημένο ορισμό από διεθνείς οργανισμούς. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει μια έκθεση για αυτό το θέμα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να βρούμε έναν ορισμό ο οποίος θα εξηγεί τι είναι η φιλοκτονία. Είναι ένας ουδέτερος ως προς το φύλλο όρος που αφορά μαζική δολοφονία ανθρώπων που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο φύλλο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε κάποιες χώρες. Και οι συνέπειες είναι μοιραίες. Είχαμε γυναικοκτονία στο παρελθόν και υπάρχουν πολλές σχετικές εκθέσεις και ψηφίσματα. Τον Οκτώβριο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εθέτησε ένα ψήφισμα για τις δολοφονίες γυναικών ε, και αφορούσε το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική και βεβαίως το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, για τη βία κατά των γυναικών και τον Απρίλιο του 2009 η Προεδρία εξέδωσε μία δήλωση και θα φτάσουμε σε κάποια δίκη για το θέμα αυτό και μετά υπήρχε μια δήλωση και διάφορα άλλα σχόλια. Προσπαθούμε να μιλήσουμε περισσότερο για την φιλοκτονία η οποία επικρατεί σε κάποιες ε, χώρες και πολιτισμούς όπως η Ινδία ή η Κίνα αλλά εμφανίζεται και στην Ευρώπη, στην Αλβανία και αλλού. Το αίτημά μου ε, ήταν να μιλήσουμε λοιπόν περισσότερο για την φιλοκτονία, δηλαδή ε, τη δολοφονία του εμβρίου. Όταν η γυναίκα διαπιστώνει ότι το βρέφος θα είναι ε, κορίτσι ή αγόρι, υπάρχει η συνήθεια σε κάποιες χώρες και επικρατούσε ο επικρατών πολιτισμός να ρίξει το παιδί αν είναι κορίτσι. Γιατί προτιμούν αγόρι για να διαιωνιστεί το όνομα και τα Και, και βεβαίως ζητήματα πρίκας και τα λοιπά και άλλα στερεότυπα και ανισότητες εις βάρος των γυναικών. Από την παιδική ηλικία, ακόμα και από την ηλικία στην οποία μένει έγκυος μια γυναίκα. Οπότε ζήτησα να μην επεκταθεί το πεδίο της έκθεσης για να μιλήσουμε για βία κατά των γυναικών ή για την έκτρωση. Δεν είναι ζήτημα έκτρωσης. Όλοι έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν αν είναι υπέρ ή κατά της ε, έκτρωσης. Ε, πρόκειται για μια έκθεση κατά της ε, δολοφονίας του εμβρίου με βάση τη διάκριση, με βάση το φύλλο και προσπαθούμε να βρούμε έναν ορισμό. Ε, προσπάθησα να επιτύχω ένα συμβιβασμό, δυστυχώς πρέπει να πω κύριε Πρόεδρε πως είχαμε πολύ λίγο χρόνο γιατί υπήρχαν τροπολογίες σε πολλές γλώσσες, είχαμε μόνο την αγγλική μετάφραση Δευτέρα βράδυ, πάρα πολύ αργά. Αν είχα άλλη μία μέρα θα μπορούσα να υποβάλω πολλές ε, συμβαστικές προτάσεις, δεν υπήρχε χρόνος. Προσπαθήσαμε λοιπόν στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και χθε το βράδυ να δούμε τον ορισμό που είχαμε μπροστά μας Και η κυρία Ζαμπόρσκα επίσης, ε, σκιοδησηγήτρια του ΕΛΚ, είχε το δικό της ορισμό που παρουσιάζεται εδώ πέρα σε μια προφορική τροπολογία στο εκτιμώντας α, τροπολογία 2, προφορική τροπολογία 2 και μετά είχα την ευκαιρία χτες στην συνεδρίαση των σκιωδών να παρουσιάσω άλλη μια συμβαστική ε, πρόταση που είχα την εντύπωση πως ε, Μα έβρισκε όλου σύμφωνου γιατί έκανα ό,τι μου ζήτησε το ΕΛΚ. Έβγαλα κάποιες λέξεις για να βρούμε μια συμβαστική λύση. Τελικά, σχεδόν μεσάνυχτα χτες το βράδυ, φαίνεται πως υπήρχε μια εναλλακτική πρόταση του ΕΛΚ και δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν ε, συμβασμό. Οπότε υποχρεωμένοι να πω πως εάν ψηφιστεί αυτό σήμερα γιατί οι σοσιαλδημοκράτες δεν θέλουν να αναβληθεί, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και θεωρούν πως πρέπει να ψηφιστεί. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν προτείνω να καταψηφίσουμε την τροπολογία 20, εκτιμώντας α, να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία 1, γιατί είναι ε, σύμβασμος ε, της ΓΚΟΕ Πρασίνων, Φιλελευθέρων και Σοσιαλδημοκρατών και ελπίζω να περάσει, γιατί είναι καλός ορισμός. Μπορώ να σας διαβάσω και τον ορισμό αν θέλετε. Αλλά θέτει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό, τότε υπάρχει μια συμβαστική τροπολογία με την υπογραφή τη δική μου των κυρίων Ρωμέβα και Γούσταυσον που βελτιώνει ελαφρώς τον αρχικό ορισμό και θα υπερψηφίσω αυτήν. Αλλά θα ήθελα να ακούσω τι έχουν να πούν οι άλλες ομάδες γιατί χθες το βράδυ είχα την εντύπωση πως ε, με μια αλλαγή εκεί πέρα μια διατύπωση θα συμφωνούσαν όλοι. Κάτι το οποίο δεν έγινε γιατί το ΕΛΚ ε, έφερε άλλο αίτημα μεσάνυχτα. Ε, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ. Μεσάνυχτα τώρα να βρούμε λύση δεν γινόταν. Αυτά είναι τα γεγονότα. Thanks a lot and... Uh, Ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο στην κυρία Σάμπορσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ την κυρία Παπαδοπούλου για το έργο της. Η δική μας ομάδα του ΕΛΚ ε, ε, ουσιαστικά ε, θεωρεί ότι αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρήσαμε ότι είναι πολύ καλό να έχουμε αυτή την έκθεση. Και αν με γνωρίζετε εδώ και καιρό, ήδη εδώ και 5-6 χρόνια, εγώ έχω τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Όμως, ήδη η εισαγωγή της κυρίας Παπαδοπούλου μας έδειχνε γιατί ξέρετε η εισαγωγή είναι ουσιαστικά σαν μια συζήτηση επί της ε, έκθεσης, δείχνει λοιπόν ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Οι μεταφράσεις έφτασαν σε μας την τελευταία στιγμή. Ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα έγινε η τελευταία τροποποίηση του καταλόγου των ψηφοφοριών. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Έτσι θα έχουμε ακόμα 15 μέρες και αυτό δεν θα επηρεάσει την ε, δουλειά μας εδώ στην Επιτροπή. Σε 15 μέρες μπορούμε να ψηφίσουμε την έκθεση και μπορώ να σας πω ότι η ομάδα του ΕΛΚ και εγώ προσωπικά θα βάλουμε τα δυνατά μας γιατί και το ΕΛΚ υποστηρίζει την έκθεση. κυρία Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στην ε, προφορική τροπολογία για το εκτιμώντας α. Εγώ την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε ένα τμήμα της παρατήρησής μου και έχει αποσύρει τρεις-τέσσερις λέξεις από το κείμενο. Όμως ε, ε, ήδη ε, για το, είχαμε συζητήσει το θέμα prenatal sex selection. Είναι αλήθεια ότι στο εκτιμώντας α υπάρχει το sex selection, αλλά σε ένα άλλο πλαίσιο και δεν υπάρχει όρος prenatal, προγεννητικός. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η δική μου πολιτική ομάδα, εγώ είμαι εκπρόσωπος αυτή τη φορά της πολιτική ομάδα και ζητά την αναβολή της ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα αίτημα να το ρυθμίσουμε αυτό το θέμα, αλλά θέλω να επενθυμίσω στους ε, βουλευτές ότι αν αυτό το θέσουμε κατά μέρος θα χάσουμε την έκθεση. Δηλαδή αυτή είναι η τελευταία μέρα που η έκθεση μπορεί να ψηφιστεί και αν δεν το κάνουμε τότε θα εξαντληθεί ο χρόνος. Έχουμε αυτή τη χρονοθυρίδα που θα χαθεί, έχουμε αυτή την ευκαιρία που θα χαθεί. Θα έχουμε λοιπόν μια έκθεση λιγότερη σε αυτή την περίοδο. Συμφωνώ με την αξιολόγηση της κυρίας Ζαμπόρσκα. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να εργαστούμε με αυτόν τον τρόπο μέσα στα μεσάνυχτα, σίγουρα. Αλλά αν δεν ψηφίσουμε σήμερα θα έχουμε πρόβλημα, να το έχετε κατά νου αυτό. Να κάνουμε έναν έλεγχο για το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας καταρχήν. Λοιπόν, αν θέλετε να ψηφίσετε σήμερα, να ψηφίσετε ναι. Αν θέλετε να ψηφίσετε σήμερα, να πατήσετε το πράσινο. Ενώ αν δεν θέλετε να ψηφίσουμε σήμερα, κόκκινο. Άρχεται η ψηφοφορία. Och voteringen är stängd. Πέρας. Λοιπόν, εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία. Πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα, λοιπόν. Ε, then I want to say something about this, uh... Και να πω κάτι ακόμα για το κτήμοντες α και την σχετική προφορική τροπολογία 1. Εστάλει πάρα πολύ αργά χθε ως συμβιβαστική τροπολογία και δυστυχώς δεν υπάρχουν κανόνες για να καθορίσουμε πόσο αργά μπορεί να στείλει κάποιος τη συμβιβαστική τροπολογία. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να αλλάξετε αυτή την προφορική τροπολογία, συμβιβαστική τροπολογία, είναι εντάξει αυτό. Αλλά νομίζω ότι το τελευταίο τρίτο τμήμα δεν μπορεί να να ανήκει σε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια νέα διατύπωση τόσο εκτενή. Επομένως, ε, η προφορική τροπολογία που θέλει η κυρία Παπαδοπούλου να την αλλάξει σε συμβαστική τροπολογία, μάλλον θα την υιοθετήσουμε μερικώς. Και θα σας πω ακριβώς ποιο είναι το τμήμα που δεν ανήκει στο συμβιβασμό. Να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Παρακαλώ, κυρία Γκαρσία Παρέση. για τις ε, τροπολογίες που παρουσίασα για την έκθεση αυτή. Κυρίως αφορούσαν ε, το θέμα της ε, φιλοκτονίας, της γυναικοκτονίας σε σχέση με τη δουλειά της κυρίας Παπαδοπούλους. Κατανοώ ότι έχει άλλο στόχο, επομένως θέλω να αποσύρω τις τροπολογίες που παρουσιάστηκαν για την έκθεση αυτή, ακούγοντας την εισαγωγή της γήτριας. Μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τι εννοείτε, γιατί έχετε πρόσφατα καταθέσει πάρα πολλές τροπολογίες, ε, δηλαδή τις ε, αποσύρετε, τι εννοείτε. Ναι, αποσύρω όλες τις τροπολογίες, λέει ο Μιλήτρια, καθώς όλες είχαν να κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα της γυναικοκτονίας. Έτσι, λοιπόν, ε, θα ήθελα οι τροπολογίες που έχω καταθέσει εγώ να μην ψηφιστούν, να αποσυρθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, αν κάνω κάποιο λάθος, να με διορθώσετε. Μάλιστα, κυρία Γκαμπριέλ. Θέλω να πω ότι όπως ε, είδαν όλοι οι συνάδελφοι ότι δεν είναι λογικό να εργαζόμαστε έτσι. Είμαστε τη στιγμή της ψηφορίας ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις ενδείξεις της κάθε ομάδες. Ενώ τώρα είμαστε ακόμη στη στάδιο να μας εξηγείτε ποιο ποιοι είναι οι συμβεσμοί, ότι εργαζόμαστε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πολύ μικρές ε, προθεσμίες ε, και στο παρελθόν είχαμε και σύγχυση μεταξύ φιλοκτονίας και γυναικοκτονίας και είδαμε με τη δεύτερη παρέμβαση ότι μέχρι την μέρα της ψηφορίας δεν έχουν ξεκαθαριστεί αυτά τα πράγματα στην έκθεση. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι αιτιολογείται το αίτημα τη πληροφορία Δεν είναι λογικό να εργαζόμαστε έτσι και η ομάδα του ΕΛΚ θέλει να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Είμαστε εντελώ ανοιχτοί. Είναι πάρα πολύ σημαντική έκθεση αυτή και το να μας δίνεται την δυνατότητα ω μέλη της Επιτροπής να καταλήξουμε σε μια έκθεση που να είναι σημαντική και συγκεκριμένη, εγώ όλο αυτό θεωρώ ότι είναι κρίμα. Και έτσι λοιπόν Αναρωτιέμαι γιατί δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τον Ιούλιο, γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη ψηφοφορία που να προβλέπεται στην εβδομάδα της 10 η Ιουλίου. Πρόεδρος, δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πρόσφατα αποφασίσαμε, ψηφίσαμε μόλις τώρα για αυτό το θέμα αποφασίστηκε ότι πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Επομένω, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον Ιούλιο και ο λόγο είναι γιατί θα χάσουμε ένα σλότ. Γιατί αν δεν ψηφίσουμε σήμερα, δεν θα είμαστε σε θέση να έχουμε την επόμενη έκθεση. Αυτά σα ενημερώνω εγώ ως πρόεδρος, αλλά ούτω ή άλλω. Ε, μπορείτε να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνουμε και εγώ θα σας ακολουθήσω. Αλλά μόλις τώρα αποφασίσετε ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Επομένως αυτό πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, τροπολογία 1. Θα προσπαθήσω να πάμε αργά, γιατί είχαμε δουλειά μέσα στη νύχτα, επομένως σας πάμε σιγά σιγά. Παρακαλώ για την τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 59, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ντεβε, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεβε ΔΕΒ2 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεβε ΔΕΒ4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεβε ΔΕΒ14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DV9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα έχουμε τις τροπολογίες 67, 68, 69, 70 που είναι ταυτόσιμες, θα τις ψηφίσουμε από κοινού, αλλά έχουμε και μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία καταρχήν. Τουλάχιστον ε, βλέπω τρει αντιρρήσει. Καταπίπτει η προφορική τροπολογία. Να ψηφίσουμε λοιπόν το αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Αποσύρεται. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο. Ωραία. Πάμε στην TV6, στην επόμενη σελίδα. Σα ευχαριστώ. Υπέρ για την TV6. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. 79, 89 είναι ταυτόσιμε. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνονται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 83 αποσύρεται, 84 το ίδιο, 85, 86, 87 ταυτόσημες, υπέρ. Κατά, εποχές, κρίνεται. 88, υπέρ. Κατά, αποχές, κρίνεται. 89, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 8, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 αποσύρεται, 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 94, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, 92. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται 94, 95, 96 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ΔΕΒΕ 11 καταπίπτει 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98, 99 καταπίπτουν όχι 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τεβεπτά τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τεβε 12 δεν ψηφίζουμε. Είναι για μη ψήφι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105, 106 καταπίπτουν. Πάμε στην 111 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, να το ελέγξουμε. Την 111. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκατόν επτά. Τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά εποχές. Πρέπει να την ελέγξουμε νομίζω την 108. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπληκτή 109 επομένω Και 110, μαλιστα dv ΔΒ3, με ψήφο 112, προφορική τροπολογία, υπάρχει αντίρρηση. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο βουλευτέ που αντιτίθεται κατά πίπτη προφορική. Σφίζουμε το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. εποχέ εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. εποχέ, εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. εποχέ εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. εποχέ εγκρίνεται. Πάμε στην 117, καταπίπτει 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 115, ψήφο 118 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕΤΑ, τμήμα 1, δεν 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 124 και 125 αποσύρονται. Δεβε 10, το τμήμα 1, 2 δεν ψηφίζεται. Πάμε στο Δεβε 10, τμήμα 2 στο 2. Υπέρ κατά εγκρίνεται 126-127 αποσύρεται πάμε στην 128 συγγνώμη 127 πολύ γρήγορα πήγα 127 υπέρ κατά Αποχές. απορρίπτεται 128 υπέρ κατά Αποχές. απορρίπτεται 129 υπέρ κατά Αποχές Συγγνώμη, να το ελέγξουμε για το 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Φέρες. Απορρίπτει. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 131. Πέρας. Απορρίπτεται. Με δύο ψήφους. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω, να ψηφίσουμε λοιπόν για την 135, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 139, 136, 137 καταπίπτουν. Πάμε στην 140 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 141, 142, 143, 144 ταυτόσημες. Κύριε Ζεμπόσκα. Συγγνώμη πρόεδρε. Αλλά οι τροπολογίες 141 ε, 142, δεν είναι ταυτοσιμε 142 διαφέρει. Ένα λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Εγώ ζήτησα να ζητήσουμε ξεχωριστά την κάθε τροπολογία. Μάλιστα. Λοιπόν, αντί να ελέγξουμε τώρα αν είναι ταυτόσιμε, όχι καλύτερα να τις ψηφίσουμε μία-μία για να είμαστε σίγουροι, εντάξει. Διαφορετικά θα καθυστερήσουμε. Να τις ψηφίσουμε όλες ξεχωριστά λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την 141 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145 καταπίπτει. Πάμε στην 146 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20. Παίρνω. Κατά. Αρχές Απορρίπτεται. Τώρα. Πάμε σε αυτό που έχουμε ως προφορική τροπολογία 1 και στον έγγραφό σας. Αλλά αυτό είναι άλλη θέση ο συμβιβασμό. Αλλά αν πρόκειται να είναι συμβιβαστική τροπολογία, δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα. Στο κείμενο τώρα ξεκινά Wonder Gender Science is Sex Neutral και μετά τελειώνει με το Lies at the Heart of Sex Selection. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε τελεία στη μέση του κειμένου κάπου λέει Where as gender based sex selection can take place. Εκεί πρέπει να βάλουμε τελεία. Μήπως ε, να το διαβάσετε, κύριε Συγήτρια, για να δούμε τι ακριβώς ε, ανήκει σε αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Παρακαλώ. Ναι, συμβαστική τροπολογία. Η τροπολογία υπογράφεται από τους ε, Παπαδοπούλου, Ρωμέβα και Γουστασόν. Λέει τα εξής. πρόκειται για έναν όρο ουδέτερος προς το φύλλο και αναφέρεται στη συστηματική και σκεμμένη δολοφονία ανθρώπων με βάση το φύλλο που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο φύλλο που είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό αλλά δεν αναφέρεται επαρκώς σε αρκετές χώρες και οι συνέπειες είναι μοιραίες. Και θα πρέπει να αναζητήσουμε τις ε, συνέπειες ε, όσον αφορά τις ε, πρακτικές επιλογές του φίλου όταν παίρνουν την μορφή της βρεφοκτονίας και εντός παρενθέσεων άλλοι όροι όπως η φιλοκτονία ή γυναικοκτονία ή φιλικτονία ε, που υπάρχουν ήδη και αναφέρονται στην ε, δολοφονία ε, γυναικών και κοριτσιών ως την κύρια έκφραση της βίας της των γυναικών. Αυτή είναι η συμβαστική πρόταση μάλιστα, την ακούσαμε, οπότε θα την ψηφίσουμε κιόλας. άλλαξε, δεν είναι πια προφορική τροπολογία, ήταν συμβαστική τροπολογία χτες το βράδυ. Άλλαξε λοιπόν συμβαστική τροπολογία. Ναι, ξέρω πως ήταν αργά, ήταν πάρα πολύ αργά. Αν θέλετε τον λόγο κυρία Λούλινγκ επί της διαδικασίας, βεβαίως. Με μικρόφωνο όμως. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, είναι προφορική τροπολογία μένα, όσο και αναφορά συμβαστική. Είναι όμως τροπολογία προφορική και όπως συμβαίνει για κάθε προφορική τροπολογία, πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε αν τη δεχόμαστε, αν είναι παραδεκτή. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κανονισμό δεν ε, υπάρχει προθεσμία για το πόσο αργά μπορεί κανείς να καταθέσει να υποβάλει συμβαστική τροπολογία. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει. Οπότε και το προηγούμενο βράδυ θεωρείται συμβαστική τροπολογία. Ναι, ναι, βεβαίως μπορεί. να το ψηφίσουμε. Ε, έχουμε και δουλειέ εδώ πέρα. Ε, γιατί υπήρχε μια συμβιβαστική τροπολογία που προτάθηκε χτες το βράδυ. Και αυτή είναι. Και αναφέρει ο κανονισμός. Ναι, ναι, φαίνεται. Άρθρο 161 του κανονισμού. Λέει τα σχετικά. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβαστική αυτή τροπολογία. Υπέρ, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε προφορική 2, 21, 22 και η 13 της ΔΕΒΕ πίπτων. Οπότε δεν έχουμε και την 20. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 αποσύρεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 αποσύρεται. 27 υπέρ. Συγγνώμη. 27 και 28 και 29 καταπίπτουν. Οπότε περνάμε στην 30. 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΔΕΒΕ 1 δεν ψηφίζεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 39 δεν ψηφίζεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε στην 45 με χωριστή ψηφοφορία και με προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις ε, για την προφορική τροπολογία ωραία θα ψηφίσουμε λοιπόν ε, μέρος πρώτο υπέρ Υπήρχε αντίρρηση. Μέρος πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε πάμε σε 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 50 προφορική τροπολογία, υπάρχει κάποια αντίρρηση, όχι, οπότε τίθεση ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 51 υπέρ, ναι, συγγνώμη, 51, 52 και 53 αποσύρονται, 54 υπέρ κατά αποχές απορριφθείτε 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ επαλήθευση της 55 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα, άρχεται η ψηφοφορία, με συγχωρείτε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4, 5, 6, 7 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 8, 9, 10, 11 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 12, 13, 14, 15 ταυτόσημες υπέρ, κατά αποχές δεκτές. Μετά προφορική τροπολογία. Έχει κάποια αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Και ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. και εγκρίνεται η έκθεση. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Σχέδιο έκθεσης. Ναι, επί της διαδικασίας κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ανακοινώσω ότι δυνάμει του κανονισμού καταθέτει εμπροθέσμους η πολιτική μου ομάδα γνώμη της μειοψηφίας.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 εγκρίνεται. Πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.